Ε, Καλώ ήρθαν οι προσκεκλημένοι μα. οι συνάδελφοι τη Επιτροπή περιβάλλοντο, Έχουμε αυτή την κοινή ακρόαση για τι νέε τεχνικέ βελτίωση. Ο κύριος Πάβελ Πότ, εκπροσωπεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς ήρθατε εσείς και τα μέλη της Επιτροπής σας. Εγώ θα κάνω την εισαγωγή στο πρώτο πάνελ και ο κύριος Πότ στο δεύτερο. Πάντως το θέμα αυτό των νέων, τεχνικών βελτίωσης είναι πολύ σημαντικό και για τις επιτροπές γιατί Έχουμε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, το θέμα των, της ποιότητας των εδαφών, του ύδατος ε, και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να τα προσεγγίζουμε όλα αυτά τα κοινά θέματα από διαφορετικές σκοπιές, τη σκοπιά των γεωργών, αλλά και τη σκοπιά του περιβάλλοντος. Σίγουρα οι νέες τεχνικές ε, βελτίωσης ε, έχουν μεγάλη σημασία για τη γεωργία ε, σε όλο τον κόσμο και σίγουρα οι γεωργοί μας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ε, πολλαπλές προκλήσεις, τις κλιματικές αλλαγές, ε, τον περιορισμό των γεωργικών εδαφών και όλο και περισσότεροι γεωργοί και επιχειρήσει ασχολούνται εντεργά με τις νέες τεχνικές βελτίωσεις. Αλλά ε, οι νέε τεχνικέ βελτίωσεις εγείρουν πολλές σημαντικές ερωτήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να, να αντιμετωπίσουμε κάποιες ε, νομικές αβεβαιότητες ε, και ε, νομικέ ανακρίβειες που υπάρχουν. Γι' αυτό διοργανώνουμε και αυτή την ακρόαση για να δούμε ε, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί και να διαμορφώσουμε και τη δική μας γνώμη για το θέμα γιατί πραγματικά το ζήτημα των νέων τεχνικών βελτίωσης εγείρει πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Θα έχουμε δύο πάνελ στην ε, δημόσια κρόση. Να καλωσορίσω καταρχήν όλους τους εμπειρογνώμονες. Ο πρώτος ε, εμπειρογνώμονας στο πρώτο πάνελ είναι ο κύριος Νίλς Λόουαρς, που είναι ο διευθυντής του Πλάντουμ, της Ένωσης Σπόρων της ε, Ολλανδίας των Κατοχωρών δεύτερος ομιλητής μας είναι ο κύριος Ζουλιά Μοντ, ε, μηχανικός στην οργάνωση επιλογή του, φρα... του γαλλικού λιμουζά και υπεύθυνο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο κέντρο Λανό στη Γαλλία για τη Φιλή λιμουζά. Καλώς ήρθατε κύριε Μόντ και εσείς. Και τρίτος ε, καλεσμένος, τρίτος εμπειρογνώμονας στο πρώτο πάνελ είναι ο κύριος Ιφ Μπερτό, που είναι διευθυντής έρευνας ε, της ΣΥΡΑ και ε, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας. Έχετε από 10 λεπτά ο καθένας. Και σας καλωσορίζω όπως είπα και προηγουμένως θερμότατα και θα σας δώσω σχεδόν σε λίγο το λόγο. Καταρχήν όμως να καλωσορίσω τους καλεσμένους κυρία Σλάιερ από την Ολλανδία. Και σίγουρα η Ένωση Plantum είναι πολύ σημαντική, ένωση σπόρο της ε, Ολλανδίας των κατοχωρών και χαίρομαι που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τα μέλη αυτής της οργάνωσης, της Ένωσης, ε, τη σημαντική αυτή δημόσια κρόαση. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Νίλς Λόουαρς, το Διευθυντή του, της Ένωσης um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι βουλευτές. Um, δεν σας αντικρίζω, αλλά ελπίζω να με βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα. Ασχολούμαι με τους ε, σπόρους ε, σε ολόκληρη τη ζωή μου. Έχω δουλέψει στην Ασία, στην Αφρική και κατόπιν στο πανεπιστήμιό μου. Έχω εκπαιδευτεί ως ε, ειδικό στους σπόρους και έχω αντιληφθεί την σημασία της δουλειάς σας. Ήταν και το αντικείμενο της, ε, του διδακτορικής μου διατριβής. Ε, μου ζητήσετε λοιπόν να μιλήσω για το πώς ε, αντιμετωπίζουμε με τα φυτά της προκλήσης κοινωνίας. Τα φυτά είναι τα πιο σημαντικά. Ο αέρας που ανασένουμε, το φαΐ το οποίο τρώμε εξαρτώνται από τα φυτά. Δεν θα υπήρχε ζωή χωρίς αυτά. Το οικοσύστημά μας επίσης αναπτύσσεται μέσα σε μέσω των φυτών και τα φυτά ουσιαστικά είναι ένα μέσο για την εξέλιξη. Αυτό το οποίο δηλαδή μπορούμε να προγραμματίσουμε μέσα στον σπόρο δεν χρειάζεται να διορθωθεί μετά. Αν υπάρχει γενετική αντίσταση στις ασθένειες των φυτών σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε αργότερα χημικές ουσίες και η γενετική αντοχή στην ξηρασία σημαίνει πιο ανθεκτικούς καρπούς ε, στην κλιματική αλλαγή. Βεβαίως αυτό χρειάζεται χρόνος. Η βελτίωση των φυτών δεν είναι κάτι το καινούριο. Ήδη έτσι ξεκίνησε η γεωργία πριν από 12.000 ε, χρόνια. Από την αρχή λοιπόν οι αγρότες ε, βελτίωναν τα φυτά, ξεκίνησαν με το να κάνουν τα ε, ζυζάνια παραγωγικά φυτά. Και έτσι έγινε το στάρι, έτσι έγιναν οι ντομάτες, οι οποίες αρχικά είχαν ξεκινήσει από ένα δηλητηριώδες είδες. Βεβαίως ε, συνεχίζεται η επιλεκτική διασταύρωση για να κάνουμε τα φυτά συνεχώς ε, όλο και πιο αποτελεσματικά. Μαθαίνουμε από την φύση μαθαίνουμε ότι τα φυτά χρειάζονται αρσενικά και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα και μετά από εκεί πέρα άρχισε ακριβώς ε, η διασταύρωση. Και βεβαίως ο Βάτσον και ο Κρίκ όταν ανακάλυψαν το DNA πρόθεσαν την κατανόησή μας στο μοριακό επίπεδο. Η εφαρμογή αυτής της γνώσης μας έφερε όλο και πιο αποτελεσματικές μεθόδους επιλογής όπως ε, πιο πρόσφατα τους μοριακούς ε, δείκτες αλλά και την μετάλλεξη, τα υβρίδια τη δεκαετία του 1920 και 30 και τώρα έχουμε την ε, στοχευμένη αναπαραγωγή και βελτίωση χρησιμοποιώντας το CRISPR-Cas9 κτλ. Κάθε φορά λοιπόν είχαμε μια σταδιακή αλλαγή που βασίζεται στην φυσική εξέλιξη. Όλοι οι αγρότες λοιπόν χρειάζονται καλούς σπόρους ανεξαρτήτως του εάν καλλιεργούμε κάτι στο μποστάνι μας ή αν είναι ένας αγρότης που καλλιεργεί βιολογικά και βεβαίως έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς σπόρων στη χώρα μου μόνο υπάρχουν 200 εταιρείες και βεβαίως κάθε φορά στο ιστορικό αυτό ταξίδι καταλαβαίναμε λίγο καλύτερα το τι κάναμε. Το μαύρο κουτί της διασταύρωσης ε, ή της ε, τυχαίας μετάλλαξης ε, των φυτών σιγά σιγά προχωρούσε και μπορούμε έτσι να προβλέψουμε το αποτέλεσμα. Οι πρόσφατες εξελίξεις λοιπόν ακολουθούν αυτήν την τάση. Όμως υπήρχε και γενετική τροποποίηση και βεβαίως εδώ πέρα προχωρήσαμε πέρα από την σταδιακή βελτίωση της επιλογής. Αναπτύχθηκαν φυτά που δεν θα μπορούσαν να έχουν ποτέ αναπτυχθεί στην φύση. Εκεί πέρα λοιπόν σωστά σταματήσαμε και είπαμε ότι υπάρχουν ζητήματα δεοντολογίας, ασφάλειας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και κατέληξαν όλα αυτά στην οδηγία 2018 ο αντίκτυπο αυτής της νομοθεσία ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η γενετική τροποποίηση τώρα εφαρμόζεται μόνο στα πιο σημαντικά φυτά, τη σόγια, το καλαμπόκι και το βαμπάκι από ελάχιστε εταιρείε που έχουν την νομική ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα. Στην Ευρώπη μόνο μία εταιρεία έχει αγορά για το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι της χωρίς κανένα ανταγωνισμό ούτε από δημοσία έρευνα, ούτε από επιχειρήσεις, ούτε καν από άλλε πολυεθνικέ. Πόσο διαφέρει η σημερινή συζήτηση και σήμερα μιλάμε για τις στοιχείες της ασφάλειας, της διοντολογίας και της εξουσίας. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σημαντικές διαφορές. Η στοχευμένη βελτίωση δεν αναπτύσσει φυτά που δεν θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί στην φύση ή μέσω της παραδοσιακής διασταύρωσης. Βεβαίως υπάρχουν ε, συνέπειες ε, οι οποίες ε, δεν θα ήταν αυτό το οποίο θέλαμε, αλλά αυτό δεν έχει οδηγήσει σε προβλήματα και η στοχευμένη διασταύρωση βεβαίω έχει σαφώς λιγότερες παρενέργειες και από την οικονομική σκοπιά. Θέλουμε μόνο οι μεγαλύτερες εταιρείες να χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους, αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό οι μέθοδοι αυτέ και ειδικά τα φυτά τα οποία προκύπτουν μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους μας. Η γεωργία πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Η νέα ΚΑΠ, την οποία αποφασίζεται αυτή τη στιγμή, αναφέρει πολύ σημαντικού στόχους. Και αναφέρω τρεις. Η βελτίωση των φυτών από μόνη της μπορεί να μην λύσει τα προβλήματα αυτά, αλλά βεβαίως μπορεί να συνεισφέρει στην μείωσή τους. Οπότε πρώτα απ' όλα έχουμε δύο αηφορία για το περιβάλλον με λιγότερους ρήπους. Έτσι με την βελτίωση έχουμε ανθεκτικότητα στις αρρώστιες. Ήδη γίνεται αυτό σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον έχει ξεκινήσει η δουλειά για να γίνουν τα φυτά πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή και επίσης να αντέχουν περισσότερο τα προϊόντα έτσι ώστε και οι μεταφορείς και οι καταναλωτές να μην χρειάζεται να πετάνε τόσα τρόφιμα. Επίσης, το ζήτημα της υψηλής ποιότητας θρεπτικών τροφίμων. Ναι, πράγματι, η απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε προϊόντα τα οποία έχουν λιγότερη γεύση και διατροφική αξία. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να δοκιμάσετε κάποιες ντομάτες που έχω φέρει να μου πείτε εάν είναι νόστιμες ή όχι. Δεν θα ήταν ωραίο να έχουμε και στάρι το οποίο δεν θα ενοχλεί όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Και άλλοι τέτοιοι στόχοι. Ε, ναι, αφήστε με να συνεχίσω. Το τρίτο θέμα. Η έρευνα και η καινοτομία να φύγει από τα εργαστήρια και να πάει στα χωράφια. Οι σπόροι είναι ένας ισχυρός μηχανισμός έτσι ώστε η επιστήμη η βαθιά μας γνώση για τις διαδικασίες εντός του φυτού να μεταφερθούν στο χωράφι με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Εγώ βλέπω και αλλιώς την ΚΑΠ. Θέλουμε να παράγουμε περισσότερες πρωτεΐνες στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να γίνει σε λιγότερες εκτάσεις γιατί έχουμε και τις πόλεις και τις υποδομές μας και θέλουμε να διαφυλάξουμε και τη φύση. Οπότε πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητά μας. Μια παραγωγή και η βελτίωση των φυτών βεβαίως από το 2000 μέχρι σήμερα έχει εισφέρει 70% της αύξησης της απόδοσης των φυτών. Και χωρίς αυτήν την αύξηση της τραματικής απόδοσης δεν θα, θα είχαμε πολύ περισσότερα προϊόντα που θα έπρεπε να εισάγουμε. Και αυτό θα σήμαινε ότι θα καταστρέφουμε γύρω στα 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα βραζιλιάνικου τροπικού δάσου. Για το μέλλον λοιπόν θέλουμε πιο ανανεώσιμε πρώτε ύλε και βεβαίως ε, να αυξηθεί και η οργανική ύλη στο έδαφο και για την υγεία του εδάφους και για τους στόχους του διοξιδίου του άνθρακα. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι όλα αυτά συνεισφέρουν και στους στόχους ε, του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε η βελτίωση είναι κάτι το οποίο είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά είναι και πάρα πολύ αργό. Γιατί όταν ε, αρχίζουμε να διασταυρώνουμε τα φυτά χρειάζονται μεταξύ 6 και 30 ετών ανάλογα με το φυτό και τον στόχο. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε και με τα κατάλληλα εργαλεία για τους βέλτιωτες ε, των σπόρων θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε πολύ πιο γρήγορα. Οπότε επαφείτε σε εσάς ε, τους νομοθέτες να αποφασίσετε ποιοι θα έχουν αυτά τα εργαλεία, το εάν θα πρέπει να επεκταθεί ο κανονισμός για τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς και σε φυτά που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί με συμβατικά μέσα πολύ αργότερα όμως. Για το εάν δηλαδή θα συνεισφέρουμε στους κοινωνικούς στόχους ή αν θα πρέπει να αναπτυχθούν και άλλη τομή τη επιστήμης για να αυξηθεί η παραγωγή πρωτεϊνών, που ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι. Αναμένω λοιπόν την σημερινή συζήτηση και βεβαίω είμαι και στην διάθεσή σας για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον κύριο Ζουλιά Μοντ από την εταιρεία για την επιλογή του, της φυλής Λιμουζά, τη βελτίωση της φυλής Λιμουζά στη Γαλλία. Ε, επίσης είναι στον πόλο του Λανό, Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και έχετε το λόγο κύριε Μόντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Ζαν που ε, μας ζήτησε να λάβουμε μέρος σε αυτή τη δημόσια κρόση μεταφέροντας τη φωνή των κτηνοτρόφων και βελτιωτών φυλής ε, λιμουζίν στη Γαλλία. Θα σας μιλήσω για τις νέες ε, τεχνικές ε, για τις θυλάζουσες αγελάδες, ταυτόχρονα λαμβάνοντας ε, υπόψη και τη βελτίωση των φυτών και αξιοποιώντα ε, την εφαρμογή των νέων τεχνικών βελτίωση και στα βοηδή. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ευρύτατο. Εγώ θα επικεντρωθώ στο θέμα του γονιδιωματικού της γονιδιωματικής τροποποίησης ή γενομικής τροποποίησης. Σε αυτές τις τεχνικές θα περιοριστώ. Καταρχήν, ε, ε, να μιλήσω ως χρήστης των νέων τεχνολογιών και όχι ως εμπειρογνώμονας της ε, ίδιας της Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το διευκρινίζω. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ε, που εργάζομαι, τον Πόλο Λανό, που είναι το αρχηγείο, τα κεντρικά γραφεία της φυλής Λιμουζίν στη Γαλλία. Βρίσκεται στην καρδιά της Γαλλίας και πρόκειται για μια, ε, ένα μοναδικό κέντρο για τις θυλάσσιες αγελάδες, γιατί συγκεντρώνουμε όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται με την γενετική επιλογή και την γενετική βελτίωση της φυλής Λιμουζίν στη Γαλλία. Και μάλιστα Ε, οι ίδιοι κτηνοτρόφοι ε, και όχι κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στη διαχείριση αυτού του πόλου. Οπότε η γενετική στις θυλάζουσες ε, αγελάδες και γενικώ στα βοηδή στη Γαλλία βρίσκεται στην κυριότητα των κτηνοτρόφων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όχι στα χέρια των μεγάλων εταιριών. Σε ό,τι αφορά τις δομές αυτού του πόλου, καταρχήν έχουμε μία μονάδα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε να έχουμε κάποια εργαλεία ε, επιλογής των μεθόδων βελτίωσης για τους κτηνοτρόφους και ασχολούμαστε κυρίως με την γονιδιωματική ε, επιλογή. Δηλαδή ε, προσπαθούμε να βρούμε στις ε, ζώνες του DNA που ε, είναι υπεύθυνε για το φαινότυπο των ζών. Δηλαδή φαινότυπος το, είναι ο, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ποσότητα του κρέατος, την ποιότητα του κρέατος και ούτω καθεξής. Και παρόλο που δεν καταλήγουμε σε γονιδιακή τροποποίηση, αυτή η μεταβατική τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι μια γέφυρα για την μεταγενέστερη γονιδιακή τροποποίηση. Δηλαδή εντοπίζουμε τις ζώνες του DNA που είναι αρμόδιες για το φαινότυπο. Στα προγράμματα επιλογής που έχουμε, βλέπετε στη διαφάνεια, στόχος μας δεν είναι να σας παρουσιάσουμε λεπτομέρειες στο πρόγραμμά μας, αλλά να δείξω ότι στηρίζεται σε 1.500 ακτινοτρόφους που επιλέγουν κάθε χρόνο 100.000 περίπου αγελάδες. Και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια γενετική πρόοδο με βάση τους στόχους επιλογής που καθορίζουν ήδη οι κτηνοτρόφοι και με μέρημνα τη διαφύλαξη της γενετικής ε, διαφορετικότητας και επικοινομορφίας. Και επαναλαμβάνω, ε, η γενετική είναι στα χέρια των κτηνοτρόφων και όχι στα χέρια των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Επίσης, το θέμα της χορήγησης διπλωμάτων ευρυστεχνίας ε, για τα ζώα, κυρίως για γενετικώς τροποποιημένα ζώα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς είμαστε υπέρ της τεχνικής του της γονιδιωματικής τροποποίησης, αλλά δεν είμαστε υπέρ της χορήγησης ε, διπλωμάτων ευρυστεχνίας σε ζώα, γιατί έτσι ε, την αφαιρούμε την ιδιοκτησία από τους ε, κτηνοτρόφους που έκαναν αυτή τη γονιδιωματική τροποποίηση και τη δίνουμε στις ιδιωτικές εταιρείε. Καταρχήν εδώ βλέπετε τις εξελίξεις τα τελευταία 40 χρόνια με τις μέσες αξίες των χαρακτηριστικών για παράδειγμα ε, ευκολία του κετού, ε, ανάπτυξη στον απογαλακτισμό, δυνατότητα άρμεγμας, μυϊκή διάπλαση, ε, οστική διάπλαση. Και μάλιστα ξεκινήσαμε με την συλλογή κάποιων στοιχείων επίδοσης στην κτηνοτροφική μονάδα και δεν ήταν πολύ, πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό γινόταν πολύ λιγότερες επιλογές ε, τη δεκαετία του 70. Μετά χρησιμοποίησαμε ε, σταθμούς αξιολόγησης ε, για να βάλουμε όλα τα ζώα στο ίδιο περιβάλλον και όχι στις φάρμες και να επιλέγουμε τα ζώα με βάση την γενετική τους αξία και όχι με βάση το περιβάλλον ή την διατροφή τους. Το 1996 το Ινστιτούτο Ίνερα μας πρότεινε ένα μέθοδο υπολογισμού, ε, μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού, ώστε να προσεγγίσουμε με πιο αξιόπιστο τρόπο τη γενετική αξία του ζώου ε, αποκλείοντας τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Οπότε βλέπετε πώς οι καμπύλες εκτενάχθηκαν στα ύψη, ανάλογα με το χαρακτήρα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τότε χρειάστηκε να αυξήσουμε τη μορφολογία και την ανάπτυξη των ζώων και αυτά πήγαν πολύ καλά. Τώρα για το θέμα της ε, διευκόλυνσης του κετού δεν είχαμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Βλέπετε την καμπύλη που ε, πηγαίνει προς τα κάτω. Αλλά ε, μετριάσαμε τα αρνητικά αποτελέσματα και με, μειώσαμε τη διευκόλυνση στον τοκετό, γιατί για, για την φιλή λιμουζίνη υπήρχαν προβλήματα, και θα διαρωτηθεί κανείς για ποιο είναι το ενδιαφέρον από τη γονιδιωματική τροποποίηση. Για δύο μορφολογικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα δεν έχει ε, νόημα, αλλά για, τον, ε, ε, για τη γραμμή τη ΜΟΒ που δεν είναι ε, κληρονομική, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνική για να έχουμε πρόοδο. Καταρχήν να δούμε ποια είναι η γενετική αρχιτεκτονική των γνωρισμάτων που επιλέγουμε. Βλέπετε καταρχήν ποιες ζώνες επιλέγουμε και δίνουμε και ονόματα σε αυτές τις ζώνες. Ε, φυσικά με, χαρακ... με ποσοτικά γνωρίσματα ε, έχουμε κάποια πολυγόνα, δηλαδή κάποιες ζώνες που δεν έχουν σημαντικά, σημαντική επίδραση. Οπότε προτιμούμε να επιλέγουμε ζώνες ε, του γονιδιώματος που έχουν ισχυρή επίδραση στο φαινότυπο. Τις ζώνες QTL όπως λέμε. Τώρα, ε, για τι θυλάζουσε αγελάδε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιε ζώνε, τέτοιε ε, θέσει ποσοτικών γνωρισμάτων, αλλά δεν τι έχουμε βρει ακόμη. Αλλά έχουμε πολλέ διαφορετικέ ερμηνείε ε, μερικού DNA. Γι' αυτό προσπαθούμε να εντοπίσουμε τι συγκεκριμένε ζώνε, συγκεκριμένε θέσει, ώστε να τι αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι γρήγορα θα έχουμε την ευκαιρία. Ε, λίγες είναι οι ζώνες αυτές, αλλά μερικές τις γνωρίζουμε και ήδη σε μερικές από αυτές έχουμε τεράστιες, ε, ε, τεράστια πρόοδο. Για παράδειγμα, για το γονίδιο που, που έχουν ζών, ε, ζώα που δεν φέρουν κέρατα. Αυτό το ακέρατο γονίδιο κατά κάποιο τρόπο προ, είναι ισχυρότερο σε σχέση με το γονίδιο που, φε, που δίνει ζώα που φέρουν κέρατα. Αυτό είναι ε, ισχυρό κατά 95% και η φιλή λιμουζά δεν έχει κέρατα γιατί η αποκεράτωση είναι με, βέβαια μια συνηθισμένη ε, τακτική που στόχο έχει να βελτιώσει την ευζοία και να μειώσει το φόρτο των κτηνοτρόφων. Η αποκεράτωση όμως είναι μια δυσάρεστη διαδικασία οπότε αν έχουμε ζώα ακέρατα ήδη βελτιώνουμε από την αρχή την κατάσταση. Οπότε αναζητήσαμε αυτό το γονίδιο, το γονίδιο που δίνει ζώα χωρίς κέρατα και βλέπετε από 100 καθαρό αίμα ε, ζώα λιμουζά έχουμε το καθαρό με 100% με την αναζήτηση του συγκεκριμένου γονιδίου που δίνει ακέρατα ζώα χρησιμοποιώντας την παρεμβολή του γονιδίου σε μια συγκεκριμένη φυλή. Ε, και τελικά το ζώο που, ε, έχουμε, που παίρνουμε έχει μόνο 50% γονίδια ε, λιμουζά, μετά το διασταυρώνουμε με ένα καθαρό αίμο, ώστε να εισάγουμε μόνο το συγκεκριμένο γονίδιο της φυλής, που στην αρχή είναι φυλή λιμουζά, αλλά στο μεταξύ τροποποιείται με την εισαγωγή αυτού του γονιδίου χωρίς ε, που δίνει ζώα κέρατα. Έτσι, με την τεχνική της γονιδιακής τροποποίησης, η πρόοδος θα είναι πολύ πιο γρήγορη. Ποια είναι τα ωφέλη αυτής της γονιδιακής ε, τροποποίησης. Καταρχήν, διατηρούμε την ε, ε, γονιδιακή πρόοδο διαφυλάσσοντας την γονιδιακή ποικιλομορφία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θέλουμε να μειώσουμε την γονιδιακή πολυμορφία Βέβαια, να ε, αναζητήσουμε το γονίδιο σε λίγους μονοτάβρους είναι σαν να ε, εξουδετερώνουμε την ποικιλομορφία τη γονίδια και κάτι που δεν ε, είναι το ζητούμενο. Σε παραγωγή ε, ε, βοηδών που είναι χρονοβόρες σε αντίθεση με άλλα ζώα όπως τα κουνέλια, με τέτοιες τεχνικές θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και το επίπεδο της παραγωγής. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα αντικαταστήσει τα παρόντα προγράμματα επιλογής. Είναι συμπληρωματικές οι δύο τεχνικές. Τώρα ως προς τα όρια που έχει η κοινωνική και πολιτική αποδοχή αυτής της μεθόδου. Αν αυτά τα τροποποιημένα ζώα απαγορευθούν στην παραγωγή και στην εμπορία στην Ευρώπη, τότε θα αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας παγκοσμίω. Γιατί το γαλλικό και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιλογής είναι παγκοσμίω γνωστά. Οπότε αν στο μέλλον σταματήσουμε την παραγωγή μας ή κάποιες εξοκοινωτικές χώρες στο μέλλον καλύψουν το χαμένο έδαφος εφαρμόζοντας αυτές τις νέες τεχνολογίες μας ξεπεράσουν και όλα, κάτι τέτοιο θα είναι καταστροφικό για την ανταγωνιστικότητά μας. Επίσης, αν δεν καταφέρουμε να υποχρεώσουμε μια παγκόσμια ιχνηλασιμότητα των τροποποιημένων ζώων, θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ιχνηλασιμότητα αν δεν κάνουμε αλληλούχηση στο ίδιο το ζώο ή τους ε, προγόνους του. υπάρχουν πολλές τεχνικές για τη γονιδιακή ε, τροποποίηση ε, ή την κλωνοποίηση ή επέμβαση στο έμβριο. Βέβαια, η τεχνική επέμβαση στο ε, έμβριο δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Καλύτερα λειτουργεί η κλωνοποίηση. Αλλά στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται η εκτροφή κλωνοποιημένων ζώων, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα. Το θέμα της κοινωνικής αποδοχής και η αποδοχή από μέρος των κτηνοτρόφων των νέων τεχνικών είναι σημαντικό ε, θέμα, αλλά ξεπερνά το αντικείμενο τη σημερινή ακρόαση. Πάντως, η πρακτική τροποποίησης γονιδιώματος συνιστά μια τεράστια καινοτομία και σημαντική πρόοδο, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των ζώων που προκύπτουν από τέτοιες τεχνικές και θα πρέπει το τροποποιημένο γονιδίωμα να είναι σταθερό από γενιά σε γενιά. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τη μεθοδολογία και γι' αυτό θα αποταθούμε στους εμπειρογνώμονες. Εν κατακλείδη, η Ένωση ε, Λιμουζίν που ε, στον πόλο του Λανό διαχειρίζεται αυτή την επιλογή στη φυλή Λιμουζέν ήταν ανέκαθεν υπέρμαχος της καινοτομίας και ε, υπέρμαχος της ε, παροχής ανταγωνιστικών εργαλείων στους κτηνοτρόφους ώστε οι κτηνοτροφικές μονάδες να είναι οικονομικά βιώσιμες. Επαναλαμβάνω όμως, χρειαζόμαστε κάποια εχέγγυα για τη μέθοδο αυτή. Άλλο θετικό σημείο είναι ότι αντιμετωπίζουμε τις κλιματικές αλλαγές και η τεχνολογία αγωνιδιωματικής τροποποίησης επιτρέπει καλύτερη και πιο ταχύ εξέλιξη των φυλών από ό,τι γίνεται σήμερα. Για παράδειγμα, έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα τσιμπούρια. Εντοπίζουμε στο DNA κάποια γονίδια που αυξάνουν την ανθεκτικότητα στα τσιμπούρια των βόηδων. Επίσης μειώνεται η θνησιμότητα λόγω της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας ε, στα τσιμπούρια. και στη πορεία της έρευνας ανακαλύπτουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά θα χρειαστούν 20-30 χρόνια για να εφαρμόσουν στις κοινοτροφικές ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ενεργοί σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την έρευνα μέχρι την εκτροφή και την επιλογή. Σίγουρα είναι πολλά υποσχόμενα αυτέ οι νέε τεχνικέ, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από την αποδοχή που θα έχουν και στο κοινό και στου κτηνοτρόφου για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα γονιδιακά τροποποιημένα ζώα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ιβμπερτό, είναι ο διευθυντής, ερευνητικός διευθυντής στο Μουσείο. Για τα σταλίες υπαρατυπίες και για ψεύδι Ε, ανάλογα με τον ορισμό που δίνει ο διαφάνειας και αποκάλυψη στοιχείων στους συμπολίτε μου και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γι' αυτό έκανα κάποια διασταύρωση στοιχείων και αυτό για να φωτίσω και τους συναδέλφους μου. Βλέπετε μια σειρά από κείμενα που είναι σημαντικό να δει κανεί ε, το δεύτερο μέρος, γιατί τα τελευταία 50 χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, μη οι τεχνικές βελτίωσεις που είναι τεχνικές ε, περιγραφικές. Καταλαβαίνουμε ότι μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών δεν υπήρχε θέμα σύγκρισης. Υπάρχει μια σειρά εμπειρογνωμόνων που λένε ότι οι τεχνικές αυτές είναι καταστροφικές ως προς τις αλλοιώσεις και τις ε, υπερβολικές αλλοιώσεις που δεν ε, μπορούσαν να προβλεφθούν. Εάν δούμε τώρα την βελτίωση των ειδών ως ε, μια εικόνα, σκεφτείτε την ιστορία αυτή ως ένα μεγάλο βόα που προσπαθούν εδώ και χρόνια, 10.000 χρόνια, να τα βελτιώσουν οι προγονείς μας από τότε. Αυτή τη στιγμή αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία 50 χρόνια σε σχέση με το σώμα αυτού του βόη είναι ένα μικρό λέπι. Ε, ένα μέρος αυτού του λεπιού, γιατί τη βελτίωση των φυτών την επιδιώκουν οι προγονεί μας τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως δεν είναι θέμα της ε, παράδοσης ε, που είχαμε ως τώρα. Επίσης βλέπουμε ποιες είναι οι απρόβλεπτες συνέπειες των τεχνικών βελτίωσης. Υπάρχουν πολλές κυρίως γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται με την ε, αλληλεπίδραση του γονιδιώματος με το επιγονιδίωμα, το επί ε, αναγράφημα, την ε, καταγραφή του γενοτύπου και του φαινοτύπου. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και ότι μόνο μερικά πετυχημένα πειράματα τελικά γίνονται γνωστά. Οι τεχνικές βελτίωσεις, τα οποία επιμολύνουν. Οπότε, όπως για τα γενετικώς τροποποιημένα που είναι ε, αποτέλεσμα διασταύρωσης, για όλες αυτές τις ε, μεταλλάξεις βλέπουμε ότι έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες και το τι αποτέλεσμα μπορεί να ε, και όλες οι υπογραφές που έχουν σχέση με αυτήν την διαδικασία όπως ε, ο συνδυασμός ε, του κάποιων μορίων μεταξύ τους, ε, το λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό, διότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της επιτάχυνσης που έχουν τις τεχνικές αυτές τα τελευταία χρόνια. Όπω είπαν και προηγούμενοι, παρά τι ε, μεταλλάξει, τι αλλοιώσει, τα τραύματα αυτά που υπάρχουν, θα υπάρξουν και κάποιε αναδιασταυρώσει για να αντιμετωπίσουν το συνδυασμό των ε, γονιδιωμάτων ή την ε, χρήση των αναδιασταυρώσεων σε περίπτωση φυτών που είναι αϊθαλοί ή που αναπαράγονται διαρκώς. Εδώ τελικά έχουμε φοβερές απώλειες από τις βάσεις δεδομένων που δεν καθαρίζονται στο γονιδίωμα των φυτών. Προ στιγμή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και γι' αυτό το λόγο, ε, παραδείγματι, κάποιοι υπεύθυνοι ε, φτιάχνουν μεγάλα θερμοκήπια, ας πούμε, ε, μεγάλες αίθουσες κλιματιζόμενες, αυτό που θα ήθελαν ε, να πετύχουν μέσα σε πολύ λίγο διάστημα σε ένα κλειστό χώρο και θα έπαιρνε δεκαετίες για την Ήπεθρο. Ε, Πάντω το γονιδίωμα των φυτών είναι φοβερά ποικιλόμορφο. Ακόμα και μεταξύ δύο ειδών καλαμποκιού, αραβοσίτου, υπάρχει η ίδια γονιδιακή απόσταση όπω μεταξύ του ανθρώπου και του πυθίκου. Όπω ε, θα διαπιστώσετε, είναι ότι όσοι ε, τις προτείνουν αυτές τις τεχνικές βελτίωσης του γονιδιώματος και του επιγονιδιώματος, χρησιμοποιούν τεχνικές προσωμείωσης ε, της βιοτεχνολογίας της δεκαετίας του 70, κάτι που καθόλου δεν απεικονίζει αυτά που γνωρίζουμε σήμερα ε, σε όλες τις ε, επιστήμες και τους κλάδους της ε, γονιδιακής. Εδώ λοιπόν με όλα αυτά τα τραύματα που έχουμε εντοπίσει πρέπει να σκεφτούμε ότι το μόνο που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι η τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί, το προϊόν που προέκυψε και η διαδικασία. Εδώ βλέπουμε να προκύπτουν τα γάματα όμικρον που είναι άγνωστα. Και εδώ βεβαίως ε, έχουμε καταλήξει στην ε, καταγραφή του Μητρώου ε, με το σύστημα καταγραφής της των δεκτυλικών αποτυπωμάτων, της κόρης του οφθαλμού, έτσι ανοιχνεύαμε το DNA. Και η διαδικασία είναι παρόμοια αυτή χρησιμοποιεί και η ΕΦΣΑ. Είναι η προσέγγιση του Μητρώου, η βιομετρική, αυτό που χρησιμοποιεί η αρχή ασφάλειας των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία επιτρέπει να πιστοποιήσουμε ότι οι μη επιθυμητές αλλαγές είναι αφυσικές, διότι κοιτάμε γονιδιακή πολυμορφία για την προστασία των φυτών και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό που πραγματικά με διασκέδασε στην ε, ε, όλη αυτή ε, η διαφιλονικία που παρακολουθώ από μακριά είναι το τι χρησιμοποιείται ε, ως επιχείρημα και η όλη επικοινωνική που μένει να θυμόμαστε τα φυσικά προϊόντα, τα παραδοσιακά, την φύση. Γιατί έγινε όλο αυτό. Διότι οι δημοσκοπήσεις στον πληθυσμό έδειξαν ότι δεν θέλει τίποτα ο πληθυσμός. Πρέπει να χρησιμοποιήσει ψαλίδια που θα κόψουν το γονιδίο μας σε συγκεκριμένα σημεία και το σύστημα αποκατάστασης του ε, και γίνεται διαμιάς. Ε, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό, διότι πρέπει να έχει προηγηθεί πολλή δουλειά. Ε, γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε υπάρχει απόλυτη εχνηλασιμότητα. Δεν μπορεί όλα αυτά να θεωρούνται φυσικά Εκτός και αν αποδεχτούμε ότι οι σημερινές κλιματικές αλλαγές είναι να προσθέτουν ε, μια σημαίνια κορνίζα στις δυσκολίες των πολιτικών να πλαισιώσουν τα θέματα αυτά, όπως έγινε λόγω χάρη με το κοινοβουλευτικό γραφείο ε, στη Γαλλία, τον Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την επιλογή των βιοτεχνολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. έχουμε μια δύσκολη κατάσταση γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερο πάνελ με επακόλουθη συζήτηση. Οπότε σας θέλω παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά στην υποβολή, στο ένα λεπτό μάλλον στην υποβολή ερωτήσεων γιατί θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο πάνελ με τη συζήτηση. Ο κύριος Άγνιο πρώτο ζήτησε το λόγο. Thank you very much. I'm... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω οι σε αυτές τεχνικές βελτίωσεις να μπορέσουν να αναπτύξουν ανοχές και όχι αντιστάσεις στην ε, αρρώστια. Πρώτη ερώτηση αυτή για τον κύριο από το Λιμουζέν. Ένα από τα προβλήματα αυτής της ράτσας είναι ότι είναι πολύ ανήσυχη, πηδάει τους φράχτες. Μπορείτε να κάνετε κάτι για να ηρεμήσει η ράτσα. Και τέλος, ε, πρέπει να το πω αυτό. Είπανε ότι κάποιοι ε, θεωρούν πως η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το φυσικό. Ναι, εγώ είμαι αυτός, θεωρώ ότι η κύκλη του ηλίου είναι κάτι το φυσικό, τα ρεύματα των ωκεανών, η περιστροφή της γης, ε, τα διαλύματα στους παγετώνες και χαίρομαι που υπάρχουν όλοι αυτοί οι φυσικοί παραγωγές. Και δεν μπορεί να με μεταπίσει κανείς ούτε καν το πράσινο λόμπι. Ναι κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους συντονιστές που δεχτήκατε την πρότασή μου για να γίνει αυτή η ακρόταση. Έχω όμως μία ερώτηση. Συχνά στο Κοινοβούλιο έχουμε μία συναισθηματική συζήτηση και όχι επιστημονική συζήτηση. Μιλάμε για τα τρόφιμα, το κλίμα, τις πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε, το τι ε, μπορούμε να κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε τα βελτιωμένα Λοιπόν, πώς μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό το οποίο θέλουμε και να καθορίσουμε τα όρια για αυτό το οποίο δεν θέλουμε. Δηλαδή, τι επιτρέπεται σε φυτά και ζώα και τι δεν επιτρέπεται για τον άνθρωπο για να μην τα, τα τσουβαλιάζουμε όλα μαζί. Αυτά και σας ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Για να ξέρετε ποιοι ακολουθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουν εξαφανιστεί εκατοντάδες εάν όχι χιλιάδες είδη. Στα αρχεία υπάρχουν διαφορά είδη που είχαν ανοχές και αντοχές. Εγώ ιδιώς καλλιεργώ 12 είδη ντομάτες στον κήπο μου και μπορείτε να έρθετε ε, να τα δοκιμάσετε. Δέχομαι οποιονδήποτε ανταγωνισμό, οι δικές μου είναι πιο νόστιμες. Στον πρώτο ομιλητή αν ήσασταν εδώ στον πρώτο μιλητή από τον FAO θα ακούγατε πως είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά πολύ η παραγωγή αρκεί να φροντίζουμε τα εδάφη μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την επιτάχυνση της βελτίωσης για να αναλύσουμε ακριβώς το γενετικό υλικό και να μην κάνουμε τυχαίες δοκιμές. Έχω πρόβλημα με την αλλαγή του γονιδιώματος και βλέπω εδώ πέρα και από τον κύριο από το την ένωση του Λιμουζέν που έχει μεγαλύτερη επαφή με τους γεωργούς που λέει δεν θέλουμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην ζωή, δεν θέλουμε να τα πάρουν αυτά οι πολυεθνικές. Το ερώτημα μου είναι πώς ε, βλέπετε να υπάρξει ακριβώς η αύξηση της απόδοσης ε, αν δεν υπάρξει κάποια εμπορική ε, σήμανση αυτών των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η σήμανση για να αποφασίζουν οι καταναλωτές εάν θέλουν να αγοράσουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέλτερ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ε, δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω και ερωτήσεις. Βεβαίως ε, το ερώτημα μου είναι αν θα μπορούσατε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου είχαμε κάποια προσαρμογή τέτοιων φυτών. Και βέβαια το δεύτερο θέμα αφορά την ε, νομοθεσία. Τα είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχει και η Κομισιόν ε, εντός αιθούς, η οποία ελπίζω πραγματικά να παρακολουθεί την, την συνεδρίαση. Ευχαριστώ τις δεκαετίες 80 και 90 του προηγούμενου αιώνα η βιομηχανία προσπάθησε ακριβώς να αλλάξει τον όρο γενετική τροπο, γενετική μετάλλαξη σε γενετική τροποποίηση. Βεβαίως αυτό δεν την βοήθησε γιατί οι καταναλωτές ξέρουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν να φάνε. Οπότε όπως και να το ονομάσουμε πρόκειται για αλλαγή ή αντικατάσταση γενετικού υλικού. Η σήμανση λοιπόν ε, και η, η χνηλασιμότητα είναι υποχρεωτικές για όλα αυτά τα υλικά. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σήμανση και θεωρώ ότι ε, θα πρέπει αυτά να καλυφθούν από την υφιστάμενη τις δύο επιτροπές ΕΜΒΗ και Άγκρη για την διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης, αλλά κάτι που είναι σκανδαλώδες σήμερα είναι να μοιράζουμε ντομάτες μιας ιδιωτικής επιχείρησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάρκεια μιας ε, ε, συνεδρίας επιτροπής. Είναι απαράδεκτο, αντιδιοντολογικό. Δεν μπορεί μια εταιρεία να κάνει προπαγάνδα με την κάλυψη ενός θεσμικού οργάνου. Παρακαλώ να σταματήσουν τέτοιες τακτικές, να απαγορεύονται τέτοιου είδους ε, ενέργειες. Είναι απαράδεκτο. Τώρα, ως προς την ουσία του θέματος για τη χρήση των νέων τεχνολογικών που ε, είναι ανθεκτικοί σε ζυζανιοκτώνα ή φυτοφάρμακα. Αυτό το στόχο έχει η γενετική τροποποίηση μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το στοχο εχει γενετικη τροποποιηση Ή έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να περιγράψουμε αυτές τις τεχνολογίες και ότι οι τεχνικοί, ε, οι ζώντες οργανισμοί ε, αναπτύσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Κύριος με ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Είναι πολύ χρήσιμη η, η δημόσια αυτή ακρόαση και σε εκμεταλλεύσει, αλλά και τις βιολογικές. Έχουμε ε, βιολογικούς γεωργούς που χρειάζονται απεγνωσμένα νέους σπόρους για βιολογικούς ε, σπόρους πατάτας, για πιο ανθεκτικά προϊόντα. Οπότε και η βιολογική ε, παραγωγή επωφελείται από τις νέες τεχνικές βελτίωσεις και τις εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό και άλλες πτυχές. Ε, επίδραση των τεχνικών στο περιβάλλον. Υπάρχει, αν υπάρχει μικρό... Δεν θα πρέπει να τα κάνουμε, να τα αναγάγουμε όλα σε ιδεολογικό ή θρησκευτικό αγώνα. Να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα και για τις νέες τεχνικές. Ο κύριος Ντενανό. Πρώτα απ' όλα σύμφωνο με τους συναδέλφους ε, έχω κάποιες ερωτήσεις για την ε, γενετική τροποποίηση θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την διάκριση μεταξύ φυσικής και μη φυσικής ε, βελτίωσης και εμένα δεν μου φαίνεται πολύ σωστό δεύτερον νέες μέθοδοι βελτίωσης. Μπορούμε να εγγυηθούμε την ελευθερία επιλογής των αγροτών. Και τρίτη ερώτηση. Αν έχετε κάποιες προτάσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική πρωτεϊνών και πρωτεϊνούχων φυτών. Κύριος Ντενανό, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δικότητα, πρέπει να σκεφτούμε την ε, βελτίωση των φυλών και των ε, σπορών. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης τι γίνεται και σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο όμως. Που... Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον για τις δύο πρώτες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να πω το εξής. Ε, το συζητάμε εδώ πέρα πάρα πολύ έντονα για αυτές τις μεθόδους ακριβώ να υπάρχει αυτή η χνηλασιμότητα. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι να είναι εμφανή. Στην αγορά με τις νέες τεχνικές βελτίωσεις. Η σχετική οδηγία διέπει ένα σύνολο τεχνικών. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Ε, φέρνουμε εδώ ή αυτό που κάνουν στην Κίνα με τα μικροχειρίδια που έχουν γίνει ζώα συντροφιάς τα οποία δεν ελέγχονται, η τεχνική και τα φυτά που προκύπτουν από αυτές τις ε, τεχνικές βελτίωσεις δεν είναι γενετικώς τροποποιημένοι οι οργανισμοί. Με συγχωρείτε εδώ, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ μπορεί να μα ε, εγγυηθεί ότι τα προϊόντα αυτά θα καταλήξουν και στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το διακύβευμα είναι αν μία νομοθεσία θα πρέπει να καλύπτει και αυτές τις νέες τεχνικές βελτίωσης. Ε, να δούμε, οι νέες τεχνικές βελτίωσης ε, περιλαμβάνουν τους ίδιους κινδύνους που είχαν και τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα, οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί. Αυτό πρώτο το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσουμε. Ο κύριος ε, ε, Μπερτό μας μίλησε για τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα τι ανεπιθύμητα αποτελέσματα υπάρχουν με τις νέες τεχνικές βελτιώσει και ποια είναι η επιρροή του στο περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα και ούτω Τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τι ανεπιθύμητα αποτελέσματα υπάρχουν με τις νέες τεχνικές βελτιώσει και ποια είναι η επιρροή του στο περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα και ούτω Γιατί σήμερα δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτών των τεχνικών σε ό,τι αφορά τα δυνητικά του αποτελέσματα. Μπορείτε να μα το διευκρινίσετε. Αυτά τα off-targets ή να επιτύχουμε τέτοια η εχνηλασιμότητα. και εσείς τι περιμένετε από την ομοθεσία και πώς θα εξασφαλίσει την εχνηλασιμότητα Voicelink. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, ο κύριος Χοίτεμα είπε ότι αλλάζουμε τη φύση προς το συμφέρον μας, προς όφελός μας. Προ το όφελος ποιο όμως, γιατί προς το παρόν η αλλαγή της φύσης φαίνεται ότι εξυπηρετεί περισσότερο ε, κάποιες ε, και δεν είναι η αλλαγή προς όφελο. Να μας δώσει μια απάντηση. Γίνεται μια περιπτωσιολογική ανάλυση των αποτελεσμάτων των γενετικών στροπημένων οργανισμών. Γίνεται περιπτωσιολογική ανάλυση της νομοθεσίας για, τα, για τους γενετικώς στροπημένους οργανισμούς όπου γίνεται στην Γερμανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Ο κύριος Χόισλιν και μετά ο κύριος Φλάναγκαν. Δικαίωμα να γνωρίζουν και πρέπει να έχει το δικαίωμα και ο καταναλωτής είναι λοιπόν ε, θεμελιώδες ε, ζήτημα. Ονειδίωμα θεωρείται σε κάθε περίπτωση κάτι το επικίνδυνο, αλλά θεωρείται κάτι το φυσιολογικό στη γεωργία. Δεν μου φαίνεται πολύ λογικό και κύριε Μπερτρόξης, μακροπρόθεσμα. Και έτσι έχουμε τελείως ε, διαφορετική κατάσταση τελικά. Ευχαριστώ. Um, it αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό αν δείτε αυτούς ε, για την συζήτηση του εδάφους, άσχετο αν τα πετάμε. Αλλά αν θέλουμε περισσότερα εδάφη, γιατί να μην μεγιστοποιήσουμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον πορεία, χωρίς να ξέρουμε τους κινδύνους. Καλό είναι το να δούμε το τι ο κύριος Μπερτό. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω εγώ, γιατί ε, απευθύνθηκαν σε μένα σε κάποιες ερωτήσεις για τις νέες τεχνικές βελτίωσης, είτε είναι το CRISPR, Cas9 ή άλλες. Έχουμε πολλές μεταλλάξεις, ε, επιμεταλλάξεις και πολλά παρεμπίπτοντα αποτελέσματα εκτός στόχου αλλά και κάποιε βλάβε. Δεν είναι κάνουμε πλήρη αλληλούχηση όλων των οργανισμών, δεν μπορούμε να έχουμε εχνηλασιμότητα. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε κάποιε προβλέψει για κάποια παρεμπίπτοντα αποτελέσματα, εκτό στόχου που μπορούν να μα επιτρέψουν να αποφύγουμε κάποια πράγματα που δεν βλέπουμε. Οι επιλάξει και ε, οι μεταλλάξει και επιμεταλλάξει μπορεί να έχουν και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που θα επεκτείνονται σε αποτελέσματα πολλά χρόνια μετά. Επίση, οι κατευθυντήριε γραμμέ δεν αρκούν. Για πολλά χρόνια είχαμε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά τώρα είναι παροχημένες. Είναι από τη δεκαετία του 70 και 80. Θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών. Ιδιαίτερα για την ε, επιγενετικότητα. Ε, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές τροποποίησεις του γονιδιώματος. Τώρα, γιατί θα πρέπει να τη θεωρήσουμε, ε, γιατί θα πρέπει να θεωρήσουμε γενετική τροποποίηση. Γιατί στην ιατρική την αποκαλούμε γενε, γονιδιωματική ή γενετική τροποποίηση. Γιατί στα φυτά να χρησιμοποιούμε άλλο ορισμό ή άλλη ονομασία. Προπέδε και, μια, και ένα δημοσίευμα ετοιμάζω με μία συνάδελφο. Θα έχετε λοιπόν πολλές λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Εγώ έκανα μία σκιαγράφηση κάποιων καταθετηριογραμμών γραμμών και πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε και αυτό κάνουν οι αρμόδιοι της επιλογής. Ε, θέλουν την, μπορούμε ε, να εντοπίσουμε τις τεχνικές και να εξασφαλίσουμε χνηλασιμότητα γιατί στους απαγόνους ε, εντοπίζουμε πολλά τέτοια γνωρίσματα. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε η χνηλάτηση αυτών των προϊόντων. Είχα πάει με άλλους τρεις υπαλλήλου στην Κίνα πρόσφατα για κάποια ε, προϊόντα που δεν επιτρέπονται να καλλιεργηθούν στην Κίνα και έφτανε σε εμά. Τώρα, 13 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να έχουμε επιτακτική ανάγκη εντόπισης ε, αυτών των ε, αυτών των κινέζικων κερασιών που ενώ απαγορεύονται στην Κίνα θα πρέπει όλα να τα δούμε επιμέρους. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μια γενική εποπτεία αυτών το προϊόντων. Γιατί ε, το βαμβάκι στην Κίνα χρησιμοποιείται το γενετικό στροποποιημένο και χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια ζωή, φυτά και δέντρα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο τι κάνουμε στη Ιαπωνία και α, ποια είναι τα αποτελέσματα σε μια καλλιέργεια, γιατί ο βαμβακοκαλλιεργητής αντί να χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα, ακριβώς ε, χάρη στα γενετικό στραπημένα βαμβάκια γλιτώνει τα φυτοφάρμακα, αλλά πλήττονται άλλε καλοί. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Απλώς ήθελα να δείξω ότι τομάτες στην αγορά ήταν λίγο άγευστες πριν από 20-30. Ότι αυτό δεν ισχύει. Όπως είπα, όλοι οι γεωργοί θέλουν καλού καλούς καλέ καλές και όλοι οι γεωργοί φύση. Η φύση δεν υπήρχε περίπτωση να βάλει 60.000 φασολιές σε ένα εκτάρι. Ε, το ίδιο και με τη βελτίωση του έως η εξέλιξη των ειδών εξαρτάται από τις μεταλλάξεις πρώτα απ' όλα και μετά από την επιλογή. Έτσι φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Είμαστε όλοι Μερικές από αυτές τις τεχνικές βελτίωσεις ακριβώς κοιτάζουν να αξιοποιήσουν τις συζήτησεις αυτέ. όμως βλέπω ότι ο Πρόεδρος θέλει να σταματήσω, οπότε θα πάψω. Θα ξεκινήσω απαντώντας για την ε, φιλή του Λιμουζάν. Φαίνεται ότι κάποιος βουλευτής ξέρει καλά το Λιμουζάν και αυτή την περιοχή και την φιλή μας. Είναι όντως άτακτη η φιλή αυτή διότι αυτό βελτιώνει και τη ζωή των κτηνοτρόφων. Είναι θέμα γενετικής γονεδιακής βελτίωσης. Άκουσα ότι τα τελευταία 40 χρόνια είχαν ήταν ε, μια φυλή δεν ε, έχει πια παρά μόνο τέσσερις τάβρους και εκατό γελάδες, είναι δύσκολο να προασπιστεί κανείς την ε, γονιδιακή της. Διότι στην Γαλλία και στην Ευρώπη κιόλας έχουμε ένα σύστημα εχνηλασμότητας των ζώων πολύ εξόπιστο. Ξέρουμε που βρίσκονται τα ζώα, μπορούμε να ελέγξουμε τις επιδόσεις του τι κάνουν τα ζώα, όλα αυτά καταγράφονται σε βάση δεδομένων και ε, μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει με τα τροποποιημένα ζώα. Βεβαίως βρισκόμαστε ακόμα σε περιματικό επίπεδο. Και μου παρετεί ομιλία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λοιπόν. Πολλές ε, ερωτήσεις υποβλήθηκαν στους καλεσμένους του πρώτου πάνελ. Φαντάζομαι θα έχουμε το... και για το δεύτερο πάνελ ε, απορίες. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ που είναι οι νέες ε, τεχνικές βελτίωσεις και το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Για το... Από το... Ο κύριος Σάρεντ Στρέγκ από το... την οργάνωση για τα διπλώματα. Στο κύριε Πρόεδρε που πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, οι νέες τεχνικές βελτίωσεις και είναι ένα θέμα όχι μόνο για μας τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά και για τους ε, ε ποικιλίε και εξάγουμε τους πόρους που παράγουμε από αυτές σε όλο τον κόσμο και μάλιστα 30% του κύκλου εργασιών μας, δηλαδή 10 ε, σπούδασα στην ε, Ολλανδία, βιοτεχνολογία και ασχολούμαι ιδιαίτερα με τις νέες τεχνικές βελτίωσης ε, και κυρίως το ε, μοιράζονται 10 μόνο εταιρείε. Οι περισσότερες ε, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είναι από τις τοπικές ανάγκες, τις κλιματικές αλλαγές και στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των πελατών. Βέβαια, τα προγράμματα βελτίωσης καταλήγουν σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Όπως συζητήθηκε και στο πρώτο πάνελ, η βελτίωση των φυτών ε, έχει μακρά και γνωστή ιστορία. Από ε, το 1866, από τους λόγους του Μέντελ για τη γενετική, είχαμε βελτίωση φυτών και μάλιστα συνεχώς ε, καταλήγουμε σε νέες ποικιλίε με διασταυρώσεις, υβριδισμό και την επιλογή των καλύτερων σπόρων. Και μάλιστα η έρευνα υψηλής τεχνολογίας είναι έρευνα ακριβίας. Χρησιμοποιούμε υβριδισμό, διασταύρωση, υποβοηθούμενοι με γενετικούς δείκτες επιλογή και γενικώ τεχνικές που εμπλουτίζονται στην πορεία του χρόνου. Βέβαια έχουν γύρει και κάποιες ανησυχίες αυτές οι νέες τεχνικές βελτίωσεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να λάβουμε υπόψη το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το τομέα. Η οδηγία 2019-2018 είναι πολύ σημαντικός. Αυτός ο ορισμός θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα. Μπορεί ο τεχνικές γε, γενετικής τροποποίησης, τεχνικές που δεν καταλήγουν σε γενετική τροποποίηση και τεχνικές γενετικής τροποποίησης όπου το προϊόν, κανονιστικό καθεστώς των νέων προϊόντων, κάτι που θα επηρεάσει και την παγκόσμια αγορά σπόρων. Και τώρα, γιατί υπάρχει επιτακτική ανάγκη του προσδιορισμού αυτού του νομοθετικού. Γιατί ε, σαν τη δική μας εταιρεία, τη Rexan ε, και άλλες εταιρείες είναι πολυεθνικές και τα προγράμματα βελτίωσή τους ε, εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο, οι πολλοί σπόρων τους γίνονται σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό, οπότε η καινοτομία είναι κινητήριος μας δύναμη. Ε, και οι ψηλές δυνατότητες που έχουμε στις τεχνικές βελτίωσεις θα πρέπει να καταλήξουν σε αξιόπιστα προϊόντα, αξιόπιστο υλικό με τη μορφή σπόρων, ώστε να συμβάλλουμε στην ε, ε παγκόσμια που προκύπτουν από νέες τεχνικές βελτίωσεις. Ε, σε άλλες περιπτώσεις ήδη είχαμε ασφάλεια δικαίου ως προς το βασικό αυτό ερώτημα. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Γεωργίας πρόσφατα δήλωσε ότι δεν ε, ε, ε, ρυθμίζει ότι πρόκειται να ρυθμίσει φυτά και βελτίωσης δεν θα θεσπιστούν νέοι κανόνες και διατάξεις. Δεύτερον, επίσης σημαντικό θέμα, το γεγονός ότι κάποιες ποικιλίε, φυτικές ποικιλίε που γίνονται από νέες τεχνικές βελτίωσης μπορούν, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ, να μην διακρίνονται από μεταλλάξεις ε, που γίνονται με γενετική τροποποίηση δεν διαφέρουν από μεταλλάξεις που γίνονται φυσικά. Για παράδειγμα, η περιόδης ε, ακτινοβολία ε, προκαλεί κάποιες μεταλλάξεις. Τέτοιες μεταλλάξεις είναι κινητήριος δύναμη της εξέλιξης, γιατί δημιουργεί μια γενετική καταλήξουν σε νέες φυτικές ποικιλίε και να προσφέρουν τα τρόφιμα του μέλλοντος. Οι νέες τεχνικές βελτιώσεις είναι πολλές, αυτή που έχει συγκεντρώσει πολύ προσοχή από κάποιες φυσιολογικές, φυσικές μεταλλάξεις ή από μεταλλάξει που γίνονται μετά από γενετική τροποποίηση. Οπότε οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν και εξασφαλίσουν σαφήνεια για το κανονιστικό καθεστώς των νέων τεχνικών βελτίωση, Επειδή οι περισσότερες νέες τεχνικές ε, και τα ε, μεταλλάξει που είναι αντικείμενο γενετική τροποποίηση, επειδή γίνεται διάκριση μεταξύ όλων αυτών, δύσκολο θα είναι να εφαρμόσουμε την οδηγία για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού σε προϊόντα που είναι αποτέλεσμα νέων τεχνικών βελτίωση. Αυτά και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να το δυνατόν και να εξασφαλίσετε μια σαφήνεια στο νομοθετικό πλαίσιο, όχι μόνο για τις εταιρείε βελτίωση φυτών, αλλά και για τους αγρότες και τους καταναλωτές της Ευρώπης που καθημερινά εξαρτώνται από τα προϊόντα μας. Ευχαριστώ. Thank you indeed. And our next speaker is Mr. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπάρτς, υπεύθυνος του Τμήματος Γενετικής Μηχανικής του Ομοσπονδιακού της Υπηρεσία Υπηρεσίας Προστασίας των Καταναλωτών και Ασφαλείας του Τροφίμου στη Γερμανία. Ευτική αρχή και ως επιστήμονας ε, που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο. Οπότε η πρώτη μου απόφαση ήταν να δώσω την τρέχουσα κατάσταση όπως ακούσαμε και από τους ομιλητές, ήδη χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική στην γεωργία, στην βιοοικονομία, στην ιατρική. Ένα αγαπημένο μου παράδειγμα είναι ότι έχουμε εμβόλια γενετικά τροποποιημένα για τις γάτες, οι οποίες ήδη έχει ανακύψει από το 2007 από την ομάδα εργασίας των κρατών μελών, όλων των κρατών μελών δηλαδή, που ετοίμασε μια τεχνική έκθεση το 2012 η οποία ακόμα επισήμως δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εάν την αναζητήσετε θα την βρείτε σε site αφόρων ΜΚΟ. Υπήρξε μια έκθεση του Κοινού Κέντρου Έρευνας ε, που δημοσιεύτηκε το 2011 και μια έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλευτικού Μηχανισμού. Περσίνη είχαμε και την ΕΦΣΑ που εξέδωσε μια γνώμοδότηση για αυτές τις τεχνολογίες και κάποια κρατημέλη που έχουν λάβει αποφάσεις για κάποιες εφαρμογές. Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ορλανδία, Ισπανία, Φινλανδία και το σημαντικότερο αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου που αναμένεται φέτος το καλοκαίρι. Αυτό είναι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα από τον Ιανουάριο φέτος και Έχουμε τώρα την ερμηνεία από την δική μας την αρχή. Αν δούμε την οδηγια 2018 που είναι βίβλος, όταν μιλάμε για την κατάταξη νέων τεχνολογιών έχουμε την κλασική γενετική τροποποίηση, έχουμε κατόπιν κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες ε, λοιπόν τροποποίηση ε, τροποποίησης ε, και βεβαίως έχουμε έναν τομέα που αυτά τα δύο αλληλεπικαλύπτονται τις νέες ε, τεχνολογίες κάποιες από αυτές ίσως και πολλές ανάλογα με την τεχνολογία με αυτήν την εισαγωγή όπου εισάγεται στο γονιδίωμα ενός οργανισμού ένα κομμάτι DNA που σαφώς εμπίπτει στον κανονισμό και ασαφές είναι αυτή τη στιγμή το κατά πόσον ε, ακριβώς αλληλεπικαλύπτονται. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το τι πρότεινε στο δικαστήριο ο Γενικός Εισαγγελέας. Ξέρω πως δεν είναι η τελική απόφαση, αλλά ίσως είναι μια ένδειξη για το προς τα που πηγαίνουμε. Λέει λοιπόν ότι έχουμε τις τεχνικές μεταλλαξιγένεσης, ε, που γίνονται είτε με ακτινοβόληση είτε με την αλλαγή, όπως είπαμε, του γονιδιώματος. Όλα αυτά οδηγούν σε έναν ε, μεταλλαγμένο οργανισμό και το κριτήριο είναι το άρθρο 2, το οποίο αφορά το εάν θα μπορούσε στην φύση να εμφανιστεί ένας τέτοιος οργανισμός και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια, δηλαδή αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην φύση, δεν είναι γενετικά τροποποιημένος οργανισμός. Εάν πληρούνται τα κριτήρια, πάμε προς τα δεξιά και πηγαίνουμε στα παραρτήματα. Και έχουμε το κριτήριο 1β1, κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή εάν πληρούνται τα κριτήρια, εάν όχι είναι ξεκάθαρα γενετικά τροποποιημένος οργανισμός, εάν ναι είναι γενετικά τροποποιημένος οργανισμός που εξαιρείται από την οδηγία. Και de facto λοιπόν έχουμε έναν ορισμό που βασίζεται σε διαδικασία και προϊόν. Επίσης πρέπει να διαβάσουμε τη γνωμοδότηση γιατί η αρχή της προφύλαξης νομίζω εκτιμάται πάρα πολύ καλά λέει εκεί πέρα ότι η αρχή της προφύλαξης δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μηδενικό κίνδυνο η ίδια η ύπαρξη του κανονισμού αυτού είναι η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και η άρνηση χρήσης νέων τεχνολογιών επίσης έχει κάποιους κινδύνους. Και τέλος, Ακόμα και αν ο νόμος περί γενετική τροποποίησης δεν ε, ισχύει για έναν οργανισμό, υπάρχουν άλλε διατάξεις που ισχύουν. Δεν ε, είμαστε δηλαδή μόνοι μα με αυτά τα φυτά ή και ζώα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για εμένα και για άλλους νομίζω από ό,τι άκουσα και από τις ερωτήσεις η καινοτομία είναι κάτι το περιπλοκό, πιο περιπλοκό από την προφύλαξη Ξεκινάμε πάνω από αριστερά, δηλαδή χρειαζόμαστε καλή ρύθμιση με όρια αλλά και ενθάρρυνση. Χρειαζόμαστε μια τεχνολογία η οποία θα είναι εφικτή. Ακούσαμε ότι σημειώνεται σημαντική πρόοδος ε, σε αυτό αλλά και από την πλευρά της οικονομίας και της οικολογίας υπάρχει ανάγκη της βιωσιμότητας και τέλος υπάρχουν οι καταναλωτές, υπάρχουν οι ανθρώπινες αξίες, πρέπει λοιπόν να είναι και επιθυμητό το προϊόν και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό από την αγορά. Να ευστήσω την προσοχή σας σε μια νέα έκθεση, ίσως και όχι τόσο νέα, που συνέταξαν πολλά γερμανικά ομοσπονδιακά όργανα το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Αξιολόγηση Κινδύνου, το Ινστιτούτο Max Χούπνερ, το Friedrich Leffler, όπου βλέπουμε πολλές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ε, όσον αφορά την ανείχνευση και ταυτοποίηση της ε, γενετικής τροποποίησης και να πω το εξής. Έχουμε κάποιες παρενέργειες, αλλά είναι σαφώς λιγότερες από την χημική βελτίωση ή την βελτίωση με ακτινοβόληση. Τελείωσα ε, γρήγορα. Ε, το βασικό μου ερώτημα λοιπόν Το βασικό ερώτημα ε, το έχω αναφέρει και σε ένα άρθρο εδώ πέρα βλέπετε στο επιστημονικό αυτό περιοδικό μας, το οποίο είναι το περιοδικό προστασία των καταναλωτών και ασφάλειας τροφίμων, εάν δηλαδή ο φόβος των δυνητικών κινδύνων των νέων μεθόδων βελτίωσης μας ε, καθιστά αδυναμούς μπροστά στις αναγκαίες αλλαγές για την βελτίωση της ζωής μας. Αυτά και ευχαριστώ ε, για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τα δύο λεπτά που δεν χρησιμοποιήσατε. Περνάμε κατευθείαν στην τελευταία ομιλήτρια η Σοφία Λακντάρ της Ένωσης Κονσόμ Ακτέρ από την Γαλλία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα μιλήσω γαλλικά και με συγχωρείτε και οι τα μου στα γαλλικά είναι, δεν είχα χρόνο να μεταφράσω. Όλοι μας, τρεις φορές τη μέρα το λιγότερο, τέσσερις ή πέντε τρώμε. Η διατροφή είναι φυσικά βασικό στοιχείο της καλής μας υγείας και της ευζοίας γενικώ. Γι' αυτό και η διατροφή είναι ένα θέμα της ε, καθημερινής πρακτικής που δημιουργεί μια τάση. Αυτό μπορεί να γίνεται μόνο με τρόπο διαφανή και ε, με απόλυτα ε, κρυβείς πληροφορίες για τη μεταλλαγή των ζώων. Μία γαλλική με κυβερνητική οργάνωση, η γιατροί του κόσμου, πριν από 10 χρόνια, είχε αποφασίσει να οργανώσει μια γαλλικη με κυβερνητικη οργανωση για αυτη του κοσμου πριν απο 10 χρονια ειχε αποφασισει να οργανωσει μια διασκεψη για την υγεία και το περιβάλλον ήταν κάτι το καινούριο την εποχή εκείνη, γιατί κανεί δεν μίλαγε ακόμη για την υγεία και το περιβάλλον σε συνδυασμό, τουλάχιστον με τρόπο ανοιχτό. Και αυτό άλλαξε λίγο τα, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Έτσι γίναμε ε, και συμμετείχα και εγώ σε αυτήν την ένωση ε, των δρόντων για την κατανάλωση. Αυτό που είναι σίγουρο βέβαια είναι ότι σήμερα και εδώ και μια δεκαετία η αύξηση της κατανάλωσης ε, βιολογικών προϊόντων ε, γνωρίζει τάση αυξητική στην Ευρώπη και στη Γαλλία και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Είναι μια τάση με διαστάσεις τεράστιες και σε όλο τον κόσμο. Η ε, υπηρεσία βιολογικών προϊόντων που είναι γαλλική υπηρεσία καταγράφει τα στοιχεία της καταναλώσεως αυτής και επιτρέπει ε, να δοθεί ο απαραίτητος χώρος σε αυτούς τους νέους καταναλωτές. Η εμπιστοσύνη στα βιολογικά προϊόντα, στις βιολογικές καλλιέργειες, με συγχωρείτε, ως ε, καταναλωτές ε, των ε, βιολογικών μπορούμε σε συνθήκες εμπιστοσύνης να αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά. Έχουμε και την εγγύηση ότι παίρνουμε προϊόντα χωρίς φυτοφάρμακα και γενετικώς τροποποιημένα. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε την κατανάλωση αυτών των προϊόντων. και η κίνηση αυτή έχει μεγάλη επιρροή και στις νέες γενιές πλέον σήμερα. Η Μεγάλες επιτυχίες από τη δεκαετία του 90 σήμερα δείχνουν ότι έχουμε καταφέρει να αγγίξουμε το κοινό. Η δική μας ένωση που δημιουργήθηκε το 2004 έχει τρεις βασικές ε, αρμοδιότητες. Πρώτον, να προφυλάξει το περιβάλλον, δεύτερον, την υγεία και τρίτον, να προωθήσει νέους τρόπους υπεύθυνη κατανάλωσης. Μέσω της διατροφής ε, προσπαθούμε να επηρεάσουμε και άλλους τρόπους κατανάλωσης όπως την ένδυση, την ε, μετακίνηση και άλλα νέα προϊόντα προϊόντα. Σκοπός μας είναι να, να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερε ηλικιακέ ομάδες από την πρώτη δημοτικού μέχρι του πολύ ηλικιωμένου και να αναδεθούν αυτά τα νέα μοντέλα κατανάλωση. Επίσης να υποστηρίξουμε και να συνοδεύσουμε, να συντροφεύσουμε αυτούς τους νέους τρόπου τρόπους κατανάλωσης και επίσης να δώσουμε επιχειρήματα στους καταναλωτές ώστε να μπορούν να προωθήσουν αυτήν τους την κατανάλωση. Επίσης το να προασπιστούμε τους καταναλωτές σημαίνει ότι προασπιζόμαστε τους εαυτούς μας κατά των τεχνικών ή των ε, παραβιάσεων που μπορεί να ε, ξεπερνούν το πεδίο ε, που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε βεβαίω ότι αυτό που μα απασχολεί σε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε και κύριοι Βουλευτέ, είναι το τι επιθυμούν οι ίδιοι καταναλωτέ για την κατανάλωσή του στην Ευρώπη. Μιλάμε για μία ένωση με 50.000 μέλη. Ε, και του αγγίξαμε με ένα ερωτηματολόγιο που απεστάλλεται τον Οκτώβριο του 2017 για του βασικού λόγου που επιλέγουν τα γελικά προϊόντα. Στο πρώτο γράφημα ε, αριστερά βλέπετε ότι 85 95% έχουν επιλέξει τα βιολογικά προϊόντα για να προστατεύσουν το περιβάλλον και την βιοπικιλότητα. 70% ε, ε, με το κίτρινο το κάνουν για λόγους ε, της πολιτικής του συνείδησης και ένα μεγάλο ποσοστό επίση, πάνω από 80% σχεδόν 90% είναι για να προσδέσει την υγεία του. Είναι τεράστιο το ποσοστό γιατί έχουμε πολλέ απαντήσει στο ερωτηματολόγιο μα. Επίση, βλέπουμε ότι ε, όσοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έχουν, ε, προέρχονται από την ύπεθρο ή το περιαστικό περιβάλλον ή το αστικό. Οι πολίτε στο αστικό περιβάλλον βλέπουμε ότι έχουν μεγαλύτερη έγνοια για το περιβάλλον από του υπόλοιπου. Επίσης, η προστασία της υγείας είναι κάτι που ε, απασχολεί ε, φοβερά τους καταναλωτές και όχι μόνο στη Γαλλία. Τα γενετικώς τροποποιημένα πάντοτε ήταν κάτι που αντιμετώπιζαν οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και μιλάμε για γενετικώς τροποποιημένα όπω ορίζονται από την Οδηγία 2001-18 και ορίζεται έτσι ένα οργανισμό πέραν του ανθρώπινου που έχει προέλθει από τρόπου μη φυσικού, με πολλαπλασιασμό ή ανασυνδυασμό σε τεχνητές συνθήκες. Έτσι θεωρούμε ότι είναι και τεχνικές βελτίωσεις ε, για τις ε, σπορές και τους γενετικώς τροποποιημένους. Θεωρούμε ως καταναλωτές ότι ε, τα όσα έχουν οριστεί στο πεδίο των βιολογικών προϊόντων ε, μας καλύπτουν και θα πρέπει να ισχύουν και για τις τεχνικές βελτίωσεις. Επίσης η οδηγία 2018 και ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις νέες τεχνικές βελτίωσεις, σε σημερινές ή μελλοντικές, είτε γίνονται όλα αυτά σε εργαστήριο είτε σε φυσικό περιβάλλον. Δεν είμαι εγώ ήδη επιστήμων και δεν θα ε, χρησιμοποιήσω επιστημονικά επιχειρήματα, λέμε καταναλώτρια. Και θα ήθελα όλα τα πειράματα που γίνονται στο εργαστήριο να μην περνάνε στο πιάτο μου. Προτού τεθούν στο ε, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και επιστοποίηση όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και μετά τη θέση στην αγορά θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον επισήμανση, ετικέτα και πλήρη ενημέρωση των καταναλωτριών και καταναλωτών. Διότι τα νέα γάματα φωμικρών πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που καλύπτουν τις ανησυχίες των ε, καταναλωτών. Όχι φυτοφάρμακα και όχι γενετικώς τροποποιημένα. Οι προτάσεις μας λοιπόν, επισήμανση σαφής που επιτρέπει του καταναλωτέ να γνωρίζουν τι καταναλώνουν, όπω με τα βιολογικά. Επίσημη απαγόρευση ε, με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων ε, για τα βιολογικά που έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα προγράμματα έρευνα, δημόσια, τα οποία να χρηματοδοτήσουν ομάδε επιστημόνων για τι νέε τεχνικέ βελτίωση. Και επίση η δουλειά των επιστημόνων να ενταχθούν στι προσπάθειε αυτέ που μπορούν να ε, επηρεάσουν μακροπρόθεσμα το περιβάλλον και την υγεία μα. Να μην υπάρξει διάδοση τέτοιων νέων οργανισμών στο περιβάλλον ανεξέλεγκτα. Τέλο, ε, και εγώ ένα σύντομο συμπερασμό ως καταναλωτρία και καταναλωτής. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι τρώμε και να έχουμε μια ετικέτα διαφανή για να περιλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις, όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο παραγωγής και την αλυσίδα ε, ε της διατροφής. Εσείς ως ε, πολιτικοί πρέπει να μα διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα διαφάνεια και προφύλαξη που πάντοτε υπερίσχυσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα θέματα τη νομοθεσία για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού είστε πλέον αρμόδιοι και πρέπει να παραμείνετε με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα ώστε να υπάρξει και η απαραίτητη κρατική συμμετοχή στα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε μάντη και σύμβιλε εδώ για να γνωρίζουμε τι ε, επιρροή θα έχουν όλα αυτά σε ό,τι τρώμε και στις μελλοντικέ γενιές. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις τεχνικές ε, του μέλλοντος από την εξή σκοπιά, να προσπαθούμε να παράγουμε χωρίς να σπαταλούμε και να μην πετάμε το 1 τέταρτο των ζώων μας από το ψυγείο. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε τον καταναλωτή, να τον προωθούμε να γίνει ε, όχι απλώς καταναλωτής βιολογικών, αλλά καταναλωτής δραστήριος των, κατανα... των βιολογικών και να μην ξεχνάμε την ιδιότητα του πολίτη και την επισητιστική κυριαρχία που θέλουμε να προφυλαχθεί και τις οποίες θεματοφύλακες είστε εσείς. Ευχαριστούμε. Thank you very much and... Ευχαριστούμε πολύ.